Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπη στις 17 Ιουνίου 2010. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 17 Ιουνίου και τα σχετικά κείμενα είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια. Όχι, τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται.